Κύριε Μέσερ Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι για τη συζήτηση αυτή τη σημερινή. Χαίρομαι που μπόρεσε να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη. Η πολιτική του ανταγωνισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είναι στοιχείο κλειδί της εσωτερικής αγοράς. Είναι σαν τον οδικό κώδικα στην κυκλοφορία την οδική. Όταν δεν τηρούμε ε, το, ε, το, πράσινο, το κόκκινο φανάρι έχουμε χάος. Έτσι είναι και εδώ με την κυρία Βεστεάρ, την ε, Επίτροπο, την ε, Δανή. Είχαμε καλή συνεργασία διότι είναι υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού. Μεγάλη χαρά. Εργάστηκα με τους σκιώδεις συγκητές των διαφόρων πολιτικών ομάδων και χαίρομαι ιδιαίτερα για του συμβιβασμούς ε, που επιτεύχθηκαν στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή και που αύριο θα ψηφιστούν στην Ολομέλεια. Υπάρχουν νέα στοιχεία που δεν είχαμε προβλέψει ε, στην πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου προηγουμένως στην, ε, ε, στην εισήγηση πρωτοβουλίας και που θα ήθελα εδώ να αναφέρω προκαταρκτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αντιμετωπίσει το κοινωνικό ντάμπινγκ. Είναι κάτι το πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι κάτι το τυχαίο, το σημειακό, είναι μια προσέγγιση οριζόντια Όποια και αν είναι η πολιτική για την οποία μιλούμε, αυτό το στοιχείο παίζει ένα ρόλο. Θα είναι ένα στοιχείο φυσικό, όπως η ισότητα ανδρών γυναικών, παραδείγματος χάρη εναέριες μεταφορές. Οι αεροπορικές πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπέστησαν μεγάλη πίεση ε, και βλέπουμε ότι οι υπάλληλοι υφίστανται αφάνταστες πιέσεις. Ε, πρόκειτο λοιπόν ε, να βρούμε μια διατύπωση που να είναι αποδεκτή για όλες τις ομάδες και ελπίζω αύριο όλοι να δεχτείτε αυτή τη διατύπωση, αυτή τη σύνταξη. Ένα άλλο στοιχείο που δεν υπήρχε στο παρελθόν είναι αυτό ε, που ονομάζουμε Leaks, τις διαρροές ως προς την πολιτική, την φορολογική που χρησιμοποιεί το Λουξεμβούργο για να ε, προσελκύσει τις μεγάλες επιχειρήσεις και να φεύγουν την μεγάλη φορολογία. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει θέση στην πολιτική ανταγωνισμού. Εξάλλου εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική ανταγωνισμού. Ελπίζω να ψηφίσουμε αύριο και ότι αυτό θα αποτελέσει βάση για μια πολιτική εναρμόνιση. Θέλουμε πάντως να υπάρχει ισότητα στους όρους. Δεν θέλουμε όλα να τα εναρμονίσουμε. Χρειαζόμαστε κρατικές ενισχύσεις, χρειαζόμαστε μια φορολογική πολιτική για τον ανταγωνισμό, αλλά θα πρέπει να είναι υγιής η πολιτική αυτή. Τρίτο στοιχείο σημαντικό για τις χώρες μας <coughs> είναι η διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων. Αν βοηθούμε τις επιχειρήσεις είναι για να βελτιώσουμε τις συνθήκες μέσα στις επιχειρήσεις και όχι για να βοηθήσουμε στην μετεγκατάσταση. Χαίρομαι που όλα αυτά τα στοιχεία αναφέρονται στην εισήγηση αυτή και χαίρομαι που σε όλους τους τομείς όπου οι πολίτες ζητούν μια προδραστική πολιτική είμαστε πάρα πολύ ακριβείς και ενδελεχείς παραδείγματος χάρη για την οδηγία απελευθέρωσης της ενεργειακής αγοράς. Δεν ωφελεί σε τίποτα να έχουμε ενεργειακή ένωση και τα πλεονεκτήματά της, εάν δεν δημιουργήσουμε τις κατάλληλες βάσεις. Το ίδιο ισχύει και για την ψηφιακή ένωση. Εξάλλου η Επιτροπή ΙΜΚΟ συνέβαλε πολύ στη συζήτηση αυτή. Και εφόσον βρισκόμαστε στην ε, ψήφιο, ψηφιακό τομέα υπάρχει ένας πρωταγωνιστής που έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο εδώ είναι η Google. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και τον κύριο Τρεμόζα ιδιαίτερα για την βοήθειά του στον τομέα αυτό και χαίρομαι που μπορέσαμε να βρούμε ένα συμβιβασμό. Θα ήθελα να τονίσω κάτι εδώ. Η εισήγηση αυτή ε, δεν είναι κατηγορίες εναντίον της Google. Αυτό που με απασχολεί είναι ότι βλέπουμε ε, διαπραγματεύσεις που ε, τραβάνε εδώ και τέσσερα χρόνια και ότι δεν έχουμε αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε την ε, Google. Δεν θέλουμε να τη στυλιτεύσουμε, αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε την κατάσταση. Πρέπει να υπάρχουν προθεσμίες για να βρούμε μια λύση. Και ελπίζω αύριο θα δεχθούμε με μεγάλη πλειοψηφία το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κυρία Μάρκα, ε, Μάρκαρετ Βεστακέρ για να απαντήσει στην παρέμβαση του κυρίου Μέσσερ Σμιτ. Uh, Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω βεβαίω τον εισηγητή, επίσης τους σκιώδεις εισηγητές και την κυρία Κάλαν, Κάλλας που έκανε την ε, γνωμοδότηση εκ μέρους της ε, Επιτροπής Εμπορίου. Θεωρώ ότι η δουλειά που έγινε εδώ είναι πολύ στέρη και ε, τονίζει τις αξίες της βάσης αυτής της εργασίας και επισημαίνει τη θέση τους για κάποιους πολύ σημαντικούς ε, τομείς όσον αφορά τις αξίες ε, και τη βάση της πολιτικής θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι τονίζεται το πόσο ο ανταγωνισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ε, έννοιας της δημοκρατίας ούτως ώστε να αποφευθεί μεγάλη συγκέντρωση του κεφαλαίου ώστε να εξασφαλίσουμε αυτοί οι οποίοι έχουν τα ταλέντα και το ζήλο να μπορέσουν να δράσουν εντός μιας ανοιχτής αγοράς. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε, όπως γίνεται στην έκθεση ότι σε εποχή κρίσης, δεν θα πρέπει να χαλαρώνουν οι κανόνες ανταγωνισμού. Αντιθέτως, θα πρέπει να διατηρήσουμε τις αγορές μας ανοιχτές, ούτως ώστε να έχουν όλοι τις σωστές ε, δίκαιες ευκαιρίες. Και όπως ε, ελέγχθη από τον εισηγητή, η πολιτική ανταγωνισμού είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να επιτευχθούν πολλοί στόχοι. Η Ενεργειακή Ένωση, η ψηφιακή ενία αγορά και η κεφαλά Έχουμε πολλέ γνώσει που μπορούμε να μοιραστούμε μεταξύ μα και αναμένω με ενδιαφέρον τη σημερινή συζήτηση και επίση, ε, όπως είπα και στην ακρόασή μου, ε, θα συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, όσον αφορά ε, σημαντικούς τομείς της προτεραιότητας. Καταρχήν την Ενεργειακή Ένωση. Οι στόχοι εδώ είναι σχετικά απλοί, ε, αυτάρκεια, ασφάλεια και φθηνός ε, και διαρκής ανεφοδιασμός. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εφαρμόσουμε την ίδια ισχύουσα νομοθεσία. Και στη συνέχεια έχουμε μια στέρεη, και έχουμε πλατφόρμα επί της οποίας να οικοδομήσουμε την Ενεργειακή Ένωση και θα πρέπει να ελέγχουμε τις ε, ενεργειακές ε, εταιρείες ούτως ώστε να μην υπάρχουν φραγμοί στην εσωτερική αγορά, ούτως ώστε να μην περιχαρακώνονται έναντι του ανταγωνισμού. Στην ε, ενιαία ψηφιακή αγορά είναι, αρκετά, είναι προφανές ότι εδώ χρειαζόμαστε μια ενιαία αγορά, γιατί μέχρι στιγμής σήμερα έχουμε εθνικές ε, αγορές και το κόστος εδώ το πληρώνουν οι καταναλωτές και οι μικρές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε ελεύθερο ανταγωνισμό και να μπορούν οι νέες τεχνολογίες ε, να φτάσουν ως τον πολίτη. Ο ανταγωνισμός μπορεί να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις ε, να φέρει μια πρόκληση ε, προς τους μεγάλους παίκτες της οικονομίας. Όσον αφορά τα... τη φορολογία, εδώ σαν εργαλείο ανταγωνισμού. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πίσω πόρτα, αλλά την κυρίω πόρτα και να αυξήσουμε τη διαφάνεια, ώστε να μην, ε, γίνεται, να μην γίνεται εκμετάλλευση της φορολογικής ε, πολιτικής, ώστε να υπάρχουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, τώρα δίνω το λόγο την εισηγήτρια από την ΙΜΚΟ, την κυρία Κάλλας. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Επίτροπο, την Επίτροπο. Έχει σημασία να λάβουμε υπόψη την ελευθερία και την ίση πρόσβαση. Ευχαριστώ επίσης τον εισηγητή για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Ως εισηγήτρια από την ΙΜΚΟ θα ήθελα να πω ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός στις δημόσιες προμήθειες, πρόσβαση ΜΜΕ, αλλά και ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς, καθώς και η ουδετερότητα του δικτύου, οδηγούν σε πραγματική καινοτομία. Ως ε, φιλελεύθεροι όμως, ε, λυπούμε γιατί προβάλλεται περισσότερη ρύθμιση από την έκθεση αυτή για το διαδίκτυο για παράδειγμα, που είναι και από τους λίγους τομείς που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Εκπροσωπούμε εκατομμύρια καταναλωτών, αλλά και όλους εκείνους που θεωρούν ότι θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη εμπιστοσύνη για να μπορέσουν να προωθήσουν το σωστό περιβάλλον για την προώθηση της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας. Χρειαζόμαστε μία αρχή υπέρ του ανταγωνισμού που να ακολουθήσει μία ενεργή πολιτική ως προς την ψηφιακή αγορά. Δεν χρειάζονται περισσότερες ρυθμίσεις και μεγαλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο, κάτι το οποίο θα είναι επιζήμιο στις επιχειρήσεις μας. Ελπίζω η Επίτροπος να συμμερίζεται αυτή την άποψη, καθώς και οι συνάδελφοι στο σώμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κυρία Κάλλας. Ο πρώτος ομιλητής εκ μέρους των πολιτικών ομάδων είναι ο κύριος ε, Λάγκεν εκ μέρους του ΕΛΚ. Ε, κύριε Επίτροπε, ε, κύριε Σεγητά, ε, η έκθεση αυτή αναφέρεται στην θητεία του κυρίου Αλμούνια και εσείς ε, κύριε Πίτροπε αντιμετωπίσετε πρώτη φορά αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει δεσμευτεί για μια οικονομική πολιτική βάση όλων των συνθήκων με την βασική αρχή μιας ανοιχτής οικονομίας ελεύθερου ανταγωνισμού. Αυτό, αυτή την αρχή θα πρέπει να την επισημαίνουμε στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων. Και η Επιτροπή έχει διευρυμένες αρμοδιότητες όσον αφορά την απαγόρευση των καρτέλ, τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων και τις ελευθερίες, την τήρηση των ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς ε, όσον αφορά την κίνηση των κεφαλαίων και των υπηρεσιών. Αυτό το οποίο λείπει ε, είναι η δημοκρατική νομιμότητα πολλών κατευθυντήριων γραμμών και κανονισμών. Αυτό είναι ε, ε, είναι κάτι το οποίο δεν βρίσκεται μέχρι στιγμή στη δικασία συναπόφασης Και αυτό συνιστά πρόβλημα στην πληθώρα των αρμοδιοτήτων που έχει η Κομισιόν. Ε, για παράδειγμα, όσον αφορά την επιβολή προστήμων προς τη Microsoft. Αυτό είναι λοιπόν ένα σοβαρό θέμα μια σοβαρή πρόκληση και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια, κατηστία του κυρίου Αλμούνια, ήταν υπερβολικά διστακτική. Έχουν οριστεί κάποια μερίδια αγορά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών αλλά για την Google δεν έγινε κάτι τέτοιο, καθυστερήθηκε για πολλά χρόνια. Ο θέμητος ανταγωνισμός επίσης αναφέρθηκε εδώ και αυτή είναι μια δύσκολη θεματολογία. Επίσης το θέμα σε ποιο βαθμό είναι οι υπεύθυνες εθνικές αρχές όσον αφορά τις ε, εθνικές ε, επιδοτήσεις. Ε, ένα παράδειγμα, όταν τα δεδομένα τα εμπιστεύτηκαν στις χώρες μέλη, και όχι σε ανεξάρτητες ε, αρχές. Είδαμε ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ο επόμενος ομιλητής ε, για τους σοσιαλιστές, ο κύριος Τσάνι, για δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μέσσερ Σμιτ και θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις εισηγητές γιατί πραγματικά η συνεργασία ήταν πολύ καλή. Είχαμε εντελώς διαφορετικές αφετηρίες, παρ' όλα αυτά έχω την αίσθηση ότι μπορέσαμε να πετύχουμε πολύ καλούς συμβιβασμούς. Ε, εκ μέρους της δικής μου πολιτικής ομάδας θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που η έκθεση αυτή επισημαίνει ε, πολύ σωστά ε, το κοινό συμφέρον και την σημασία των ε, υπηρεσιών για τον πολίτη και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Εσωτερική Αγορά, την Επιτροπή ΙΜΚΟ για το γεγονό ότι τόνισε εδώ τη σημασία τη ψηφιακή αγορά. Γιατί πιστεύουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μέσω τη καινοτομία στην Ευρώπη. Επίση, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για το γεγονό ότι η έκθεση αυτή Ε, μας ε, εξοικειώνει με τις κοινωνικές διαστάσεις του θέματος. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι λυπηρό ε, το γεγονός ότι το ΕΛΚ θέλει να εξοβελήσει αυτές τις κοινωνικές πτυχές από την έκθεση. Αυτό για μας είναι απαράδεκτο. τα, κοινωνικές διαστάσεις θα πρέπει να παραμείνουν στην έκθεση. Ε, το σημείο 85 μπορεί να παραμεινθεί. Εδώ πρόκειται για την ε, απελευθέρωση των ε, σειροδρομικών συγκοινωνιών. Οι σοσιαλιστές λοιπόν δεν μπορούν να υποστηρίξουν εδώ αυτή την φιλελεύθερη πολιτική. Ε, και επίσης θεωρούμε το γεγονός ότι στο σημείο 45 απευθύν, ε, ονομάζεται μια συγκεκριμένη εταιρεία. Επόμενος ομιλητής εκ μέρους των φιλελευθέρων, ο κύριος ε, Κρόπαρτσικ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μέσερ Σμιτ για αυτόν την εισήγηση που είναι πολύ υψηλής ποιότητας. Ο ανταγωνισμός, η ανταγωνιστικότητα είναι στοιχεία ουσιώδη για την ανάπτυξη της Ευρώπης και έχει επιπτώσεις πάνω στις τιμές, κυρίως τιμή της ενέργειας και σύνεπώς στις δυνατότητες ανάπτυξης. Εδώ Έχουμε ένα πρόβλημα που τίθεται στην Ευρώπη, διότι συγκρίνουμε την τιμή της ενέργειας στην Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Εδώ είναι δύο φορές ψηλότερες οι τιμές. Οι τιμές του αερίου ε, πολλαπλασιάστηκαν επί 2,5 σε σχέση με την Αμερική. Αλλά υπάρχουν χώρες όπως η δική μου, η Πολωνία, όπου η τιμή του αερίου είναι πέντε φορές ανώτερη από την τιμή του αερίου στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ένα πραγματικό φρένο στην ανάπτυξη που εμβαθύνει στην ε, οικονομική κρίση της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Και τώρα μιλάμε για κλιματική πολιτική αυτή η νέα ιδεολογία που προβάλλουμε και αυτό αφήνει λίγη θέση στον ανταγωνισμό και στην ανταγωνιστικότητα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανταγωνιστικότητα ευρωπαϊκή μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Τερμόζε Μπαλσέλς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο ανταγωνισμός είναι ένας τομέας όπου η Ευρώπη μπορεί πραγματικά να καταπολεμήσει τις ολιγοπολιστικές πρακτικές. Πιστεύω ότι ο κύριος Μόρτεν Μέσσερ Σμίτ πραγματικά τα κατάφερε πάρα πολύ καλά και διαπραγματεύτηκε σωστά με όλους τους σκιώδεις για να έχουμε αυτή την τελικά καλή έκθεση στην ΕΚΟΝ είχαμε 51 ψήφους υπέρ και μόνο 2 κατά. Ελπίζω λοιπόν αύριο να υπάρχει ευρία πλειοψηφία υπερψήφισης για να αποστείλουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα προς την Επιτροπή. Κυρία Φέσταγκερ, εάν θέλουμε να φτάσουμε σε μία νέα ρύθμιση, θα πρέπει το μηχανισμός αντιτράστ ε, να δράσει τάχιστα. Ε, ως προς τη Google και τη συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα με όλους τους ενάγοντες και τους εναγόμενους, ε, αντιμετωπίσαμε το ζήτημα, αλλά ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος. Πιστεύω ότι στην περίπτωση της ε, πρακτικής αντιτράστ και της αγωγής κατά της ε, Google, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μερικοί δεν έχουν ε, πρόβλημα να εκφραστούν δημόσια, άλλοι όμως Άλλοι φοβούνται τον αποκλεισμό από την Google και έτσι δεν ε, μιλούν ελεύθερα. Πολλά θύματα αυτής της πρακτικής από την Αμερική μας είπαν πως αποκλείστηκαν από την Google αρκετές ημέρες με πολύ σοβαρή οικονομική επίπτωση για αυτούς. Εγώ δεν αντιτάσσομαι στην Google ή οποιαδήποτε άλλη ε, επιχείρηση αμερικανικής προέλευσης, αλλά είμαι κατά του μονοπωλίου. Η Google έχει 90, κατέχει το 90% ε, της πρόσβασης στο διαδίκτυο στην Ευρώπη. Η προτιμησιακή πρακτική της Google δεν είναι σωστή πρακτική γιατί δεν, είναι και, δεν χρησιμοποιεί και τα καταλληλότερα μέσα υπέρ των καταναλωτών. Θα αντιδράσει μόνο εάν υπάρξει χρηματική ποινή. Ε, κυρία Φεστάκερ, θα προβάλλετε αντιρρήσεις στην περίπτωση αντιτράστ κατά της Google. Αν θέλετε να είσαστε αξιόπιστοι, μόνο αντιδρώντας θα το καταφέρετε. Υπάρχει μία μπλε κάρτα για σας. Κύριε ε, Τρεμόζα, η Μπαρσέλς, δέχεστε την μπλε κάρτα. Κύριε Herr Φοντσούλικερ, για 30 δευτερόλεπτα. Uh, you put the microphone on, please. Παρακαλώ, ανοίξτε το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο εάν συμφωνεί με τη συμπερίληψη της, ε, του κειμένου σχετικά με την Google. συμφωνείτε, με την συμπερίληψη σε αυτή την έκθεση. Συμφωνείτε ότι υπάρχουν προσωπικές επιθέσεις κατά της Google. Και δεν, δεν είναι θέμα φορολόγησης. Εγώ δεν ζητώ να γίνει φορολογηθή, θα ήθελα να γίνει φορολόγηση. Θα πρέπει να υπάρχει ίση πρόσβαση στην Αμερική υπάρχει Yahoo η οποία μπορεί να ανταγωνιστεί την Google. Δεν ισχύει όμως ε, στην Ευρώπη κάτι τέτοιο γιατί πολλές επιχειρήσεις πλήττονται από την κακή πρακτική της Google και αν δεν κάνουμε κάτι τα επόμενα χρόνια θα απαρίσταται στην αγορά μόνο η Google. Δεν είναι θέμα ε, φορολόγησης, αν σας κατάλαβα καλά, είναι θέμα ίσης πρόσβασης στην αγορά. Όπως ξέρετε, κατά της ε, Microsoft ε, επιβλήθηκαν ε, χρηματικές κυρώσεις το 2002, 2004, 2007 και 2009. Γιατί δεν έγινε κάτι τέτοιο κατά της Google. Επόμενη ομιλήτρια είναι για 1,5 λεπτό η κυρία Λόπεθ Μπερμέχο εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Α εξολογήσουμε τα θετικά στοιχεία αυτή τη έκθεση. Ας θεωρήσουμε ότι διατυπώνει σημαντικές κριτικές και προτεραιότητες. Την στιγμή πρέπει να δοθεί ένας νέος προσανατολισμός στην πολιτική του ανταγωνισμού καταγγέλλοντας την εκμετάλλευση κατά των μικρών καλλιεργητών και καταδικάζοντας τις υπερβολικές επιδοτήσεις ε, στις τράπεζες και ε, στριλτεύοντα το κοινωνικό ντάμπινγκ. Παρ' όλα αυτά έχουμε επιφυλάξει για κάποια θέματα τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση όπως για παράδειγμα τη σημασία να ληφθεί υπόψη ο σκοπός ενός υψηλού επίπεδου απασχόλησης όπως το προβλέπουν οι συνθήκες. Η έκθεση αυτή θα έπρεπε να καταγγείλει το γεγονός ότι η πολιτική ανταγωνισμού ε, δεν θα πρέπει να είναι το εργαλείο μέσω του οποίου ε, καταστρέφονται οι δημόσιες ε, υπηρεσίες ε, η Επιτροπή ε, με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην ε, καταστροφή των θέσεων απασχόλησης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδίω σε χώρες όπως η Ισπανία. Εμείς έχουμε υποβάλει κάποιες τροπολογίε στο Κοινοβούλιο γιατί θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στους Ευρωπαίους να γνωρίσουν κατά πόσο ε, ε, οι μεγάλες ε, πολιτικές ομάδες δίδουν προτεραιότητα στις απασχόληση ή όχι αλλά η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη. Η πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να προστατεύει, προστατεύει τις δημόσιες υπηρεσίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους έναντι των ε, καταχρήσεων ε, των ε, μεγάλων ομίλων. Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ρεϊμό εκ μέρους των Πρασίνων για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ πολύ ε, αξιότιμη κυρία Πίτροπε, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Μέσσερ Σμιτ, ο οποίος ε, έκανε μια σημαντική, ένα σημαντικό έργο και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις γιατί ε, πρόκειται για μια εδώ δίκαια διαπραγμάτευση με ένα καλό αποτέλεσμα. Θα ήθελα να επισημάνω τρία σημεία τα οποία σημαντικά, θα είναι σημαντικά και πιο σημαντικά ακόμα για το μέλλον από ό,τι στο παρελθόν όταν συντάχθηκε η έκθεση του 2013. Το πρώτο είναι ότι ε, θα πρέπει να ελέγχεται η επιθετική φορολογική πολιτική ε, σε μια συγκυρία όπου ε, το, ε, τέθηκε το θέμα των Lux Leaks. Ίσως θα έπρεπε να σχηματιστεί μια ειδική επιτροπή και όχι μια απλή εξεταστική επιτροπή όσον αφορά ε, τι επιθετικέ ε, μορφέ ε, ανταγωνισμού. Τώρα, όσον αφορά την ιδιωτικότητα του δικτύου, η έκθεση τονίζει ότι είναι, έχει μεγάλη σημασία να μην υπάρχουν διακρίσει όσον αφορά τη διακίνηση δεδομένων στο ίντερνετ. Και αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ιδιαίτερα σχέση με την Google και είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν εφόσον δημιουργούμε ένα δίκτυο όπου για πολλά χρήματα γίνονται πολλές ε, αγορές. Όταν ο συνάδελφος κύριο Έτιγκερ ε, χαρακτήρισε τους υπερασπιστές της οδεδρότητας του δικτύου ως Ταλιμπάν, αυτό ήταν μια πρόγευση ε, για μια πολιτική κατεύθυνση που δεν θα οδεύει τα επόμενα χρόνια προς μια ουδετερότητα του δικτύου. Και θα ήθελα να το αποθείτε εσείς κυρία Επίτροπε. Το τρίτο σημείο είναι ότι λέμε ότι οι ανανόσιμες ε, πηγές ενέργειας θα πρέπει να προωθηθούν και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το στοιχείο της βιωσιμότητας. Πώς αυτό είναι συμβατό με μια πρόθεση ή με μια έγκριση της ε, προώθησης για ε, εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας. Πρόκειται για μια μαζική στρέβλωση του ανταγωνισμού που ενέκρινε ο προκάτοχός σας, κύριος Αλμούνια. Και εδώ θα πρέπει να κινηθούμε αποφασιστικά και σε πολιτικό επίπεδο. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος εμιλητής είναι ο κύριος Στίβεν Βούλφ ε, για δύο λεπτά, δύο μισή λεπτά. Ευχαριστώ. Η Ευρώπη πεθαίνει. Ε, τα άτομα αγωνίζονται. Οι πολίτες, ως όλη αυτή την ωραία Ήπειρο υπάρχουν οικογένειες που δύσκολα επιβιώνουν, ανεργία, τα παιδιά τους που φεύγουν, προσπαθούν να φτιάξουν τη ζωή τους σε αυτόν τον κόσμο ο ανταγωνισμός είναι ουσιαστικό μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για, να, για αυτούς που προσπαθούν να βρουν εργασία για να έχουν αρκετά χρήματα στη τσέπη τους για να πληρώσουν λογαριασμούς αερίου, ηλεκτρισμού και να θρέψουν τις οικογένειές τους. Όταν βλέπουμε λοιπόν μια εισήγηση ε, που ενός ε, εισηγητού ε, του κύριου Μέσσερ Σμιτ που δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα σε αυτήν την Βουλή. Θα υπάρχουν ε, πάντοτε τέτοιες εισηγήσει ε, που θα ε, πέφτουν σε αυτιά που δεν ακούνε, διότι στο τέλος της, τέλος της γραφής υπάρχουν εδώ κανόνες, κανόνες για τις επιχειρήσεις, αλλά οι επιχειρήσεις έχουν την εξουσία την επιρροή και έχουν πρόσβαση στους επιτρόπους, στους βουλευτές. Τους βλέπω εδώ σε αυτό το κτίριο και στις Βρυξέλλες όπου έχουν πρόσβαση στους ευρωβουλευτές και τους υποβάλλουν ιδέες, κανόνες, κανονισμούς για να υπάρχουν μεγάλα εμπόδια πρόσβασης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενθαρρύνεται όχι ο καπιταλισμός, αλλά η συντεχνική προσέγγιση ε, κερδίζουν πάρα πολλοί εκατομμύρια σε μπόνους ε, εις βάρος αυτών που προσπαθούν να επιβιώσουν. Είναι ένας τόπος επικίνδυνος όπου ο ανταγωνισμός αποτυγχάνει και καμιά εισήγηση σαν κι αυτή δεν θα επιτύχει το στόχο που θέλουμε, δηλαδή να ανακουφίσουμε ε, την, τους πολίτες οι οποίοι υποφέρουν στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Βούλφ. Έχετε ένα, μια μπλε κάρτα από τον κύριο Ιάκοφτσίτς. Για 30 δευτερόλεπτα παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Όταν μιλάτε, συμφωνώ ότι ότι οι άνθρωποι που προσπαθούν να επιβιώσουν και αγωνίζονται, όταν τους βλέπετε δεν βάζετε το χέρι στη τσέπη. Και εσείς μπορείτε να επηρεαστείτε ε, ως ευρωβουλευτής ή αποφασίζετε μόνος σας. Υπάρχουν πάρα πολλά λόμπι εδώ τριγύρω, αλλά εγώ αποφασίζω πάντοτε για τον εαυτό μου. Δεν με επηρεάζουν αυτά τα λόμπι. Αυτή ήταν η ερώτηση. Βεβαίως, ε, χαίρομαι που ελεύθερα αποφασίζετε εσείς και εγώ ελεύθερα αποφασίζω, αλλά αυτό που έχω δει εδώ στο Κοινοβούλιο, είδα ότι μεγάλα κόμματα όπως το ΕΛΚΑ και οι σοσιαλιστές πιστεύουν, ε, ψηφίζουν on block. Είναι η ελίτ του κόμματος η οποία αποφασίζει και επηρεάζεται από τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους εθνικούς πολιτευτές. Έχετε ελευθερία για τον εαυτό σας, αλλά όχι ελευθερία μέσα στο κόμμα σας. Ποια για 1,5 λεπτό η κυρία Κάπελ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Ε, ο ανταγωνισμός ε, είναι κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη και δύο ε, βασικοί παράμετροι όπου ε, και εδώ η κατάσταση στην Ευρώπη δεν είναι ιδιαίτερα ρόδινη. Υπάρχει μεγάλη μείωση της ανταγωνιστικότητας και έχει διπλάσια ποσοστά ανεργίας από ό,τι στη ΣΥΠΑ. Ε, έχουν χαθεί 6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας το περασμένο έτος, ενώ στις ΗΠΑ μόνο 1 εκατομμύριο. Οι τιμές της ενέργειας όσον αφορά το φυσικό αέριο είναι διπλάσεις από ό,τι στις ΗΠΑ ή στις Ινδίες η, ε, η επίσης τα φορολογικά βάρη είναι πολύ υψηλότερα από τις ΗΠΑ και κατά 100% υψηλότερα από ό,τι στην Ιαπωνία. Και ε, επίσης στον τομέα της έρευνας υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα, 100 εκατομμύρια, 100 ε, δις, ανά έτος. Η... Γι' αυτό η έκθεση νομίζω ότι επισημαίνει ορισμένα σημαντικά σημεία, δηλαδή στρατηγικές ε, προτεραιότητες για αυτή τη θητεία, δηλαδή ε, ξεκάθαρα και θεμετή κανόνες ανταγωνισμού, τήρηση αρχής επιχωρητικότητας, σεβασμός ε, στις εθνικές αποφάσεις, ε, ξεκάθαρα κανόνες ε, για τα καρτέλ, αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές επιδοτήσεις. μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε έχουμε μια σωστή πολιτική ανταγωνισμού η οποία θα επιφέρει πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές. Η επόμενη μιλήτρια είναι η κυρία Έστερ Ντελάνκε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ επίσης την Επίτροπο για την παρουσία της. Βεβαίως θα πρέπει να συμβάλλει ο ανταγωνισμός σε μια δίκαιη οικονομία όπου οι κανόνες του παιχνιδιού να είναι ίσοι για τις επιχειρήσεις και όπου προστατεύονται οι καταναλωτές. Θα πρέπει να διατηρήσουμε την πίεση. Βλέπουμε ότι συχνά τα κράτη-μέλη σε περίοδο οικονομικών ε, δυσκολιών δίνουν κρατικές ενισχύσεις ε, και ορθώνουν εμπόδιο. Ε, χαίρομαι που έχουμε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μεριμνά. Οι πρώτοι που υποφέρουν από την αποχώρηση με ενός κράτους από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ωφελούνται από την εσωτερική αγορά. Η ψηφιακή αγορά θα πρέπει να εγγυάται την ισότητα, την δικαιοσύνη και να προλαμβάνει τον κατατεμαχισμό τα κρατημέλη θεωρούν σημαντικότερα τα μεγάλα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων και όχι την δίκαιη και πρόσβαση των πολιτών στο διαδίκτυο. Άλλο σημείο σημαντικό είναι η νέα οικονομία της μοιρασιάς, της ανταλλαγής. Εάν παραδείγματος χάρη παίρνω ένα ταξί Uber σε ένα κράτος μέλος, είμαι παράνομος ενώ σε άλλα κράτη είμαι νόμιμος και αλλού είναι γκρίζα ζώνη. Εδώ πρέπει να εξαγάγουμε συμπεράσματα. Θα πρέπει να αποφύγουμε αυτού του είδους ε, το χάος. Ο καλός ανταγωνισμός ε, είναι καλός, αλλά για να μπορεί να υποφεληθεί η κοινωνία θα πρέπει να επαγρυπνεί η Κομίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ η Ανελίζε Ντότς για 1,5 λεπτά. Σε ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Επίτροπο που παρίσταται εδώ. Πολλές φορές λέγεται ότι η ανταγωνιστικότητα θα οδηγήσει σε ίση πρόσβαση των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και τη χώρα προέλευσης. Άρα ε, αναγνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει ίση πρόσβαση τη στιγμή που πολλές επιχειρήσεις επιθετικά δεν καταβάλουν τους φόρους τους. Το LuxLeaks ε, δείχνει ότι σε ορισμένες χώρες οι επιχειρήσεις ε, καταβάλουν φόρους κοντά στο μηδέν μετά από διμερείς συμφωνίες με τεχνητά μέσα. Άρα ο ανταγωνισμός εδώ είναι σαν αγώνα 100 μέτρων και χρησιμοποιώντας άνισα μέσα, δηλαδή ο ένας να χρησιμοποιεί τα πόδια του και ο άλλος ένα αυτοκίνητο της Φόρμουλας 1. Άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο ανταγωνισμός και η απελευθέρωση αγοράς δεν είναι πάντα η σωστή λύση. Έχει σημασία ο τομέας της υγείας, η εκπαίδευση ή σε άλλους τομείς που δεν απέδωσαν οι επιχειρήσεις. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για ίση πρόσβαση όταν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και θα πρέπει οι κυβερνήσεις να αντιδράσουν έναντι των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει να προωθήσουμε την πράσινη ενέργεια γιατί δεν έχει νόημα να έχουμε ίση πρόσβαση στην αγορά αν το, το επίπεδο πρόσβασης είναι 10 μέτρα κάτω από, το, από τη γη. Μπλε κάρτα από την κυρία Άτκινσον. Τη δέχεστε, κυρία Άτκινσον, για 30 δευτερόλεπτα με μικρόφωνο. Δηλαδή τι κάνετε ε, στην ουσία ε, υποστηρίζετε τον Γιούγκερ ο οποίος θέλει να ενώσει πάντα. Εδώ μιλάμε για το TTIP. Μιλήσαμε για την ελευθερία του τύπου και ούτω καθεξής. Εσείς θεωρείτε στην ουσία ότι, ότι υφίσταται ισότητα. Με συγχωρείτε, είμαι κρυωμένη και δεν μπορώ να μιλήσω όπως θέλω. Εσείς υποστηρίζετε την Guardian. Θεωρείτε ότι υπάρχει πραγματικά ελεύθερος τύπος ή Guardian υποστηρίζει θέσεις που δεν είναι σωστές. Χαίρομαι που προβάλλετε αυτές τις θέσεις. Θα ήθελα να πω ότι ίσως υπάρχει μια σύγχυση. Το Κοινοβούλιο έχει προβάλει αυτή την έκθεση, δεν είναι έκθεση της Κομισιόν. Άρα ακούγεται η φωνή του Κοινοβουλίου για θέματα ανταγωνισμού. Εγώ έχω επισκεφθεί τις ΜΜΕ και τις επισκέπτομαι συχνά στην εκλογική μου περιφέρεια και φοβούνται τις πολυεθνικές οι οποίες ε, μεταφέρονται σε φορολογικούς ε, παραδείσους για να μην πληρώνουν φόρους. Ελπίζω να αλλάξετε την πολιτική σας. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Πέτεσεν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσω στην ιδρική μου γλώσσα. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή για μια πραγματικά πολύ καλή έκθεση. Η πολιτική ανταγωνισμού είναι ένας από τους βασικούς τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματικά καθοριστικός ε, τομέας και είναι σημαντικός και για τη νέα Επιτροπή και για την κυρία Φέσταγκερ. Η πολιτική ανταγωνισμού είναι ένας από τους πολλούς τομείς όπου η συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θετική και επιφέρει απτά ωφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και είναι θετικό το γεγονός ότι ο εισηγητής λέει ξεκάθαρα ότι η Κομισιόν θα πρέπει να έχει περισσότερες αρμοδιότητες έναν των χωρών μελών. Και θεωρώ επίσης θετικό το γεγονός ότι ο εισηγητής τονίζει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να έχει τα οικονομικά μέσα ούτως ώστε να μπορεί πραγματικά να υλοποιήσει αυτά τα πολύ σημαντικά της καθήκοντα. Επίσης είναι θετικό το γεγονό ότι ο εισηγητής τονίζει το ρόλο του Κοινοβουλίου και λέει ότι θα πρέπει να έχει περισσότερες ε, αρμοδιότητες το, το Κοινοβούλιο γιατί θα πρέπει να συνεχίσει αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα το οποίο διαπιστώνεται αυτή τη στιγμή. Η Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να έχει περισσότερα ε, οικονομικά μέσα και το Κοινοβούλιο περισσότερε αρμοδιότητε. Αυτό σημαίνει περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι λιγότερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίω αυτή είναι μια αλλαγή στη στάση του εισηγητή. Το γεγονός ότι λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη συνεργασία. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν. Ο επόμενο ομιλητή είναι ο κύριος Μάρκο Βάλι για 1,5 λεπτό. Άκουσα ορισμένε παρεμβάσεις από συναδέλφους και θεωρώ ότι πολύ συχνά το κοινοβούλιο νομοθετεί σωστά αλλά τι γίνεται μετά. Η εκτελεστική αρχή, δηλαδή το Συμβούλιο και η Επιτροπή που θα πρέπει να εφαρμόσουν σωστά οδηγίες, ε, δεν ακούν το Κοινοβούλιο. Αναρωτιέμαι γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα Γιούνκερ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ε, προέβησε φορολογικό ντάμπινγκ υπέρ της χώρας του για 15 χρόνια, ο οποίος θα μπορούσε αύριο να προβάλλει κάτι το αντίστοιχο, γιατί έχει όλα τα μέσα. Δηλαδή η Επιτροπή σε ποιους θα δώσει συμβουλές. Τι παράδειγμα αποτελεί. Το Κοινοβούλιο εργάζεται πολύ καλά, αλλά δυστυχώς το Συμβούλιο και η Επιτροπή ε, που ορίζονται από τα λόμπι στην ουσία δεν μπορούν παρά να προωθήσουν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Και βλέπουμε ότι οι πολίτες είναι αυτοί που ζουν τις συνέπειες με την ανεργία, με, την, με τον αθέμητο ανταγωνισμό, όπου οι πολιεθνικές έχουν φορολογική έδρα εκεί που τους συμφέρει. Θα πρέπει κάτι να κάνετε γι' αυτό, διαφορετικά θα επανέλθουμε στον προστατευτισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενο ομιλητή είναι ο κύριο Μάρκο Φέρμπερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο ανταγωνισμό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της, του οικονομικού μας συστήματος. Γι' αυτό είναι ορθό ότι από την εποχή της συνθήκης της Ρώμης έχουμε μια υπηρεσία ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία μεριμνά ούτω ώστε ο ανταγωνισμός εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι θεμητός. Ε, και αυτό είναι και το δικό σας καθήκον κυρία Φέσταγκερ ε, τώρα και ε, πραγματικά σας εύχομαι καλή τύχη όταν το ζητούμενο είναι να διατυπώσετε τους κανόνες του παιχνιδιού και να μεριμνήσετε ούτε ώστε αυτοί οι κανόνες του παιχνιδιού να γίνονται σεβαστοί από όλους τους παράγοντες της αγοράς. Αυτό έχουμε να αναμένουμε από μια σωστή πολιτική ανταγωνισμού. Έχουμε πολύ μεγάλες προκλήσεις για παράδειγμα όσον αφορά το φορολογικό δίκαιο. Έχουμε συστήσει μια ειδική επιτροπή και χαίρομαι, χαιρόμαστε που η επιτροπή έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ελέγχου ε, σε σχέση με ε, κάποιες παραδιάσεις εκ μέρους των χωρών μελών. Ε, σε μια ψηφιακή αγορά δεν είναι πάντα σαφές ποιοι κανόνες του παιχνιδιού θα πρέπει να τηρούνται και θεωρώ ότι αυτή είναι μια μεγάλη ευθύνη και μεγάλη πρόκληση. Επίσης θα πρέπει να μεριμνήσουμε ούτως ώστε να μην αποδυναμώσουμε την Ευρώπη με έναν εσφαλμένα κατανοούμενο ανταγωνισμό. Ε, δεν θα πρέπει να αποδυναμωθεί η Ευρώπη μέσω των ε, κανόνων του ανταγωνισμού και θα μπορούσαμε εδώ να αναφέρουμε τις ε, ενέργειες συγκοινωνίες ή τις τηλεπικοινωνίες. Επίσης θα πρέπει να δούμε το θέμα της απασχόλησης και το λαμβάνει υπόψη αυτή η έκθεση. Γι' αυτό εύχομαι ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της όλες αυτές τις προτάσεις της έκθεσης. Η κυρία Αλέζια. Οι πολιτικοί ανταγωνισμού αποτελούν απαράβατες αξίες για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Αποτελούν ένα αναγκαίο μέσο για να αρθούν τα προσκόμματα στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, προσώπων, αγαθών και εμπορευμάτων. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι σε πολλούς τομείς υπάρχουν ε, πολλά προσκόμματα που δεν επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία μιας ε, ε, εσωτερικής αγοράς που είναι δυναμική και καινοτόμος, επιτρέποντας τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θα ήθελα να τονίσω το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα τελευταία χρόνια σε αυτό το τομέα και θεωρώ ότι τα σχέδια ανταγωνισμού θα πρέπει να εγκρίνονται σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και αναφέρομαι σε μία προέκταση ή επέκταση της διαδικασίας της συναπόφασης για να ενισχύσουμε τη δημοκρατική νομιμότητα. Το δημοκρατικό έλλειμμα είναι απαράδεκτο και θα ήθελα να αρθούν τα προσκόμματα στον τομέα του ανταγωνισμού. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός αν δεν υπάρχει διαφάνεια. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πρακτικές και τις φορολογικές συμφωνίες μεταξύ των κρατών που προβάλλει η Επιτροπή. Ευχαριστούμε πολύ επόμενος ομιλητής για δύο λεπτά ο κύριος Τόλογιαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υποστηρίζω πλήρως την έκθεση αυτή που ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει τις περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων ως προς την κρατική βοήθεια και τις φοροαπαλλαγές σε ορισμένες πολυεθνικές, ιδιαίτερα σε κράτη-μέλη. Ξέρω ότι η Επιτροπή ασχολείται με αυτό το ζήτημα και αναμένουμε τα συμπεράσματα. Θα ήθελα επίσης να λάβουμε υπόψη τις ε, πολύ διαφορετικές τιμές για τα ίδια ε, σκευάσματα, φαρμακευτικά σκευάσματα τόσο μεγάλες ε, διαφορές δείχνουν ε, καταχρηστικές ε, πρακτικές και σε επίπεδο παρασκευαστών και διανομέων. Αυτές οι μεγάλες διαφορές δείχνουν ότι η αγορά είναι κατακαιρματισμένη στον τομέα των φαρμακευτικών σκευασμάτων. Γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με αυτό το θέμα των φαρμάκων στην Ευρώπη για να εντοπίσει αγορές που κατέχουν δεσπόζουσα θέση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις καταχρήσεις αυτές. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής για 1,5 λεπτό, ο κύριος Κόφωτ. Øh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρειάζεται ελεύθερος ανταγωνισμός ε, δίκαιος για να επωφελείται ο καταναλωτής κυρίως ε, για την κινητή τηλεφωνία και για την ηλεκτρονική ψηφιακή αγορά. Σε άρθρο του Financial Times βλέπουμε ότι μας περιμένουν πολλές συγχωνεύσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να κατανοήσει ότι ότι για να εγκρίνει αυτές τις συγχωνεύσεις πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα ο καταναλωτής. Υπάρχουν στην Δανία ε, δύο εταιρείες που θέλουν να συγχωνευτούν. Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη την κατάσταση. Οι δύο αυτές επιχειρήσεις οι δανικές τι ποσοστό αγοράς μπορούν να έχουν ε, προτού να θεωρηθεί η θέση του ως δεσπόζουσα. Είναι κάτι το ουσιώδες. Δεν πρέπει να υπάρχει αύξηση της τιμής για τον καταναλωτή. Το δέχεστε αυτό ως στοιχείο βάσης. Ευχαριστώ τον κύριο Μέσερ Σπίτα για την εξαίρετη και ενδιαφέρουσα εισήγησή του και για την φιλική προσέγγιση. Συγχαρητήρια κύριε Μεσερσίτ. Ε, θέλετε περισσότερη εξουσία για ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω ε, τι θέλετε να πείτε με όλα αυτά κύριε Μέσερσμιτ, αλλά πάντως σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Γεώργιος Κίρτσος για δύο λεπτά παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, εντάξει θεωρώ ότι όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει τέλεια αγορά και πρέπει να υπάρχουν παρεμβάσεις για να περιοριστούν οι δυσλειτουργίες. θεωρώ ότι και η έκθεση του κυρίου Μέσσερσμιτ αλλά και η επίτροπος κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. θα ήθελα να σας πω σαν έλληνας ευρωβουλευτής ότι η διάστρωση της εσωτερικής αγοράς παίζει τεράστιο ρόλο στο τελικό οικονομικό αποτέλεσμα αλλά βέβαια δεν είναι όλα αρμοδιότητας της ευρωπαϊκής ένωσης πρέπει και οι κυβερνήσεις πρέπει και οι ίδιες οι κοινωνίες να ενδιαφερθούν. θεωρώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών ένας από τους λόγους που η ελλάδα δεν κατάφερε να βγει από το πρόγραμμα προσαρμογής τόσο καλά τόσο γρήγορα και με την επιτυχία που είχαν η ιρλανδία και η πορτογαλία που είχαν τα δικά τους προγράμματα ήταν τα προβλήματα στη διάρθρωση της εσωτερικής αγοράς. δηλαδή γίνανε πολλές θυσίες έπεσαν τα ημερομίσθια αλλά διατηρήθηκε ο πληθωρισμός σε ένα επίπεδο 2,5% για το 2010-2014 παρά το γεγονός ότι το ονομαστικό κόστος εργασίας μειώθηκε γύρω στο 12% και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν έπεσε 20%. Επομένως έχει τεράστια σημασία το πώς λειτουργεί κάθε οικονομία, το πώς περιορίζουμε τις δυσλειτουργίες της. το θέμα λοιπόν είναι αν από τις σωστές πολιτικές πρωτοβουλίες που θα πάρουμε θα, γίνουμε, θα καταφέρουμε να γίνουμε συγκεκριμένοι. για παράδειγμα γιατί το ρωσικό φυσικό αέριο που εισάγεται στην ελλάδα είναι από τα ακριβότερα στην ευρωπαϊκή ένωση; γιατί η μείωση του κόστους ενέργειας δεν φαίνεται στα τιμολόγια της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. αν καταφέρουμε και λύσουμε αυτά τα συγκεκριμένα νομίζω θα πάμε πολύ καλύτερα. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενο ομιλητή ε, για 1,5 λεπτό, ο κύριο Φρουντσούλητσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πολύ με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για την εισήγηση αυτή. Θα ήθελα να τονίσω ε, το αποτέλεσμα για τις δημόσιες υπηρεσίες που πρέπει να υπάγονται σε πολιτική ανταγωνισμού, τη δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να έχουν καλές δημόσιες ε, υπηρεσίες είναι κάτι το κρίσιμο ε, για την ομάδα μας των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Με τις τροπολογίες που υπέβαλα υποστήριξαν έναν μεγαλύτερο ρόλο του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση της πολιτικής ανταγωνισμού του ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια της αγοράς, η σταθερότητα και η ανάπτυξη. Ε, διαμέσου του, της εισήγησης αυτής μπορούμε να επιτύχουμε ουσιώδεις στόχους όπως να εξασφαλίσουμε ε, την, τον δίκαιο ανταγωνισμό ε, να οι υπηρεσίες ε, γενικού οικονομικού ενδιαφέροντες να υπάγονται ε, στους νόμους του ανταγωνισμού, να έχουμε αντιμονοπολιακή πολιτική, να να καταργήσουμε τις ενισχύσεις στις τράπεζες και φόρους που είναι παράνομοι, αλλά δεν, δεν ξέρω με την Google τι πρέπει να γίνει, αλλά υποστηρίζω εφόσον η ιδέα της εισήγηση είναι γενική κανόνας, ε, προτείνω να υιοθετηθεί η εισήγηση αυτή στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τον κύριο Ντέιβιτ Κάσα για δύο λεπτά. Ναι, θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας τον εισηγητή για τις προσπάθειές του Νομίζω ότι είναι πολύ ισορροπημένη η εισήγηση. Βεβαίως το θέμα του ανταγωνισμού είναι σημαντικός καταλήτης για την προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης ε, και της σταθερότητας. Το 2013 η έκθεση της Επιτροπής ε, ήθελε να δώσει περισσότερη ισχύ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διότι υποφέρει αυτός ο τομέας της οικονομίας και έχει πληγεί από τις συνθήκες στην ευρωπαϊκή αγορά. Ωστόσο, ίσως έχουν ανακτηθεί κάπως οι απώλειες, έχουν έχουμε ορισμένα διδάγματα σχετικά με, τους, με τις δημόσιες συμβάσεις, τους διαγωνισμούς, αλλά τέτοιος ε, ανταγωνισμός υγιής ε, πρέπει να επιτευχθεί με κανόνες, χωρίς την Επιτροπή δεν θα είναι οι δυνατότητες αυτές πιο προσιτές στις μικρομεσαίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να ετοιμάσει κατευθυντήριες γραμμές σαφής για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές για την νέα νομοθεσία, για τον ανταγωνισμό, για δυνατότητες καλύτερες για τις μικρομεσαίες και να μην έχει αποκλειστικά συμβάσεις που αποτρέπουν την είσοδο στην αγορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη ομελήτρια για δύο λεπτά, η κυρία Ντανούτα Ζασκοβιέτσκα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Αναμφίβολα η πολιτική του ανταγωνισμού είναι στοιχείο κλειδί της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς. Αν δεν δράσουμε αρκετά σε κοινοτικό επίπεδο μπορεί να υπάρχουν ε, εμπόδια και ίσως εμπορική πόλεμη μεταξύ των κρατών μελών και θα υποφέρουν οι καταναλωτές και το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τα νέα μέτρα της Κομισιόν. Να θυμηθούμε ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα κονδύλια για να ενισχύσουν τη θέση τους σε αγορά. Το τελευταίο έτος μας έδειξε τα προβλήματα των φορολογικών παραδείσων και την πολιτική ορισμένων κρατών. Η υπόθεση LuxLeaks μας έδειξε ότι οι κράτη θέλουν να προσελκύσουν επενδυτές και τροποποιούν το φορολογικό δίκαιο και έτσι ορισμένες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από βαριά φορολογία. Πολλές επιχειρήσεις επωφελήθηκαν από το Λουξεμβούργο, επιχειρήσεις οι οποίες είχαν κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Θα πρέπει να τονίσουμε λοιπόν τη σημασία της φορολογικής πολιτικής. Συμφωνώ ότι η διαφάνεια του φορολογικού δικαίου είναι στοιχείο σημαντικό του ανταγωνισμού και η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να έχει εργαλεία για να μπορεί να ανοιχνεύει αυτές τις κακοήθεις πρακτικές ε, στην εσωτερική αγορά έχουμε θέμα ανταγωνισμού, δεν αναφέρθηκε στην έκθεση. Έχουμε πληροφορίες ότι η τιμή ε, του ρωσικού αερίου διαφέρει από κράτος σε κράτος. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια πραγματική, ένα πραγματικό ανταγωνισμό ανάμεσα σε επιχειρήσεις αν ορισμένοι πληρώνουν 308 δολάρια για το αέριο και άλλοι 20% περισσότερο. Η τιμή αυτή δεν απορρέει από αντικειμενικές συνθήκες και εξαρτάται από την καλή θέληση της πολιτικής του Κρεμλίνου και ορισμένοι μιλάνε για κοινωνικό ντάμπινγκ χωρίς να μιλούν για ενεργειακό ντάμπινγκ όταν είχαμε την συζήτηση για την Ενεργειακή Ένωση. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μονό για 1,5 λεπτό. Μπορούμε να πούμε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού απέτυχε γιατί αν εξαφανίστηκαν ορισμένα μονοπόλια είναι για να προωθήσουν τα συμφέροντα σε ιδιωτικές εταιρείες. Ιδιωτικοποίησεις δηλαδή με βάση το σχέδιο Juncker, ιδιαίτερα στο τομέα των μεταφορών και της ενέργειας. Ο τραπεζικός τομέας που δέχτηκε δύο ε, δις μέσα σε ένα χρόνο δεν προέβαλε τίποτα. Η δικαιοσύνη κατακεραυνώνεται, δεν έχει καταφέρει τίποτα. Το βλέπουμε και στην περίπτωση της Google. Επίσης, οι δημόσιες προμήθειες δεν λειτουργούν καλά, ούτε το δίκτυο διανομής. Δεν μπορεί ένα κυρίαρχο ε, κράτος, δηλαδή, να προβάλλει μία πολιτική οικονομικού προγραμματισμού. Η SNCF χρειάστηκε ε, στην ουσία να δώσει πίσω 400 δις ευρώ διότι δεν μπόρασε ε, να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της έναντι του Βελγίου. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να μην κινούμαστε κατά των συμφερόντων των λαών. Catch the Eye. Θα δεχτώ έναν ομιλητή αναπολιτική ομάδα και όχι ομιλητές που ήδη έλαβαν το λόγο σήμερα το απόγευμα. Η κυρία Ρωμάνα Τόμιτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι η πολιτική ανταγωνισμού είναι, έχει τεράστια σημασία αν θέλουμε να αναζωογονήσουμε τις οικονομίες μας. Ειδικά σήμερα όπου αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις όπως ε, εμπορικές συμφωνίες με άλλες χώρες και θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας ε, στην πιο σημαντική εξ αυτών μεταξύ ΕΠΑ ΕΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική του ανταγωνισμού ε, είναι το μόνο εργαλείο προστασίας των καταναλωτών ούτω ώστε να οικοδομήσουμε ένα έντιμο περιβάλλον για όλες τις εταιρείε, ακόμα και τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πάντοτε είναι θύματα των αλλαγών στην οικονομία. Χαίρομαι που η Επιτροπή αναλαμβάνει ενεργό ρόλο ε, στον έλεγχο των τεκτενόμενων στην οικονομία και αναμένω με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μαρία Καμίνε για ένα λεπτό. Σίγουρα θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την ευχαρίστησή μου για την έκθεση αυτή, αλλά θα ήθελα να θίξω το εξής ερώτημα προς την Επίτροπο. Χρειαζόμαστε μια πολιτική ανταγωνισμού, αλλά σωστού ανταγωνισμού. Δεν ξέρω κατά πόσο έχετε σκεφτεί κάτι συγκεκριμένο σε δύο κατευθύνσεις. Πολιτικές που αφορούν την αντιμετώπιση των ΜΜΕ, γιατί εγώ ήμουν επιχειρηματίας και είδα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπήρχε σωστός ανταγωνισμός μεταξύ ΜΜΕ και μεγάλων πολυεθνικών. Επίσης, ξέρετε τι σημαίνει η είσοδος μη ευρωπαϊκών χωρών στην ευρωπαϊκή αγορά, γιατί έχουμε πολλά προϊόντα που δεν ελέγχουμε. Αν αυτοί οι δύο τομείς, σε αυτούς τους δύο τομείς υπάρχει έλεγχος, τότε θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την πολιτική ανταγωνισμού. Για ένα λεπτό, κύριο κύριος Άγγελ Τσαμπάσκι. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μέσερ Σμιτ για την πολύ ισορροπημένη εργασία του με πολύ ακρίβεια απέδωσε μεγάλη σημασία στις μικρομεσές επιχειρήσεις που πρέπει να προστατευθούν κατά του ανταγωνισμού των μεγάλων επιχειρήσεων διότι παρέχουν ε, απασχόληση σε 65% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι περισσότερες μικρομεσαίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν ε, και να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό των μεγάλων. Υπάρχουν ορισμένες αδυναμίες στην εισήγηση, αλλά δεν είναι και τόσο σημαντικές. Στην Βουλγαρία έχουμε επιτόκια μέχρι 50% για τα δάνεια και αυτό πρέπει να το προσέξουμε σχετικά με άλλα στοιχεία όπως ε, το κοινωνικό dumping ε, νομίζω ότι το λάβατε υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο κύριος Ιβανιός Φίτς για ένα λεπτό. Ναι. Η ελεύθερος ανταγωνισμός είναι σημαντικός για την οικονομία μας, αλλά σε αυτήν την εισήγηση είναι σαφές ότι η περισσότερη Ευρώπη σε αυτούς τους τομείς δεν ξέρω αν είναι καλύτερη για μας, διότι έχουμε προβλήματα ανταγωνισμού στον ενεργειακό, ε, ενεργειακή αγορά και στην ψηφιακή αγορά. Είπε συνάδελφος για το θέμα της Google και τη θέση της Google στην αγορά. Έχουμε μια ψηφιακή αγορά και η ελευθερία η ψηφιακή στην Ευρώπη πρέπει να είναι από τις σημαντικές ελευθερίες και έχουμε εδώ μονοπόλιο. Θα πρέπει να πάρουμε μακροπρόθεσμα μέτρα, ιδαλλιώς η κατάσταση δεν θα είναι καλή για την οικονομία μου. Ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Φερέρο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ε, η ελεύθερο, ο ελεύθερος ανταγωνισμός επέβαλε την απελευθέρωση πολλών τομέων της οικονομίας. Μας έλεγαν ότι όλοι θα κέρδισαν. Είδαμε τα αποτελέσματα στον τομέα του ηλεκτρισμού είδαμε ότι έπρεπε οι επιχειρήσεις και οι οικογένειες να καταβάλουν μεγαλύτερο αντίκτυμο. Αντίτιμο, ενώ τα κέρδη ήταν πολύ μεγαλύτερα για τις επιχειρήσεις. Στις μεταφορές η απελευθέρωση οδηγεί σε μονοπόλια. Έχουμε 6-7 επιχειρήσεις σε αυτό το τομέα. Επίσης, υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού στον τομέα της γεωργίας εξαιτίας της ΚΑΠ και δημιουργούν, δημιουργούμε παρεμβατισμό από τα κράτη εκεί όπου μας συμφέρει, δηλαδή επιλεκτικό ε, παρεμβατισμό. Τώρα κυρία Επίτροπος, κυρία Φέστακερ, έχει το λόγο. Καταρχήν θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την συζήτηση αυτή. Πιστεύω ότι έδειξε το βάθος και την δέσμευση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφόσον όταν το ζητούμενο είναι η πολιτική ανταγωνισμού και οι κανόνες που απορρέουν από τη συνθήκη. Εκτίμησα πάρα πολύ τα όσα είπε ο κ. Ε, Λάγκεν λέγοντας ότι ε, βάσει της συνθήκης δεν υπάρχει συναπόφαση με αυτό το κοινοβούλιο εγώ θα ήθελα να πω ότι όσο έχουμε αυτή τη συνθήκη ε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο αλλά θα συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο και ε, βεβαίως όταν το ζητούμενο είναι να προχωρήσουμε πιο μακριά ε, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Όπως είπε ε, κατά δεύτερο λόγο ο κύριος Πέτερσεν θα πρέπει να συνεργαστούμε πολύ στενά με τις εθνικές αρχές γιατί μόνο έτσι μπορούμε να λύσουμε θέματα τα οποία αλλιώς δεν θα μπορούσαν να λυθούν. Ε, για παράδειγμα, στον αφορά το τομέα των τροφίμων. Επίσης, οι εθνικές αρχές ε, έχουν τα δεδειγμένα εργαλεία στη διάθεσή τους. Επίσης, ε, κατά πόσο το, η πολιτική ανταγωνισμού μπορεί να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα δικά τους ε, ταλέντα για να μπορέσουν να μπουν στην αγορά. Θεωρώ ότι αυτό είναι σημαντικό σημείο γιατί ε, φωτίζει ένα από τους βασικούς στόχους της ε, πολιτικής ανταγωνισμού που είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Τώρα, όσον αφορά τις τιμές των ε, φαρμάκων και τις διαφορές εδώ, ε, η προηγούμενη Επιτροπή έκανε έναν ε, έλεγχο σε σχέση με τους κανόνες στον τομέα αυτό οι διαφορές τιμών ίσως οφείλονται στις διαφορές μεταξύ των χωρών ε, μελών όσον αφορά τις επιδοτήσεις των φαρμάκων. Βεβαίως ε, θα ε, παρακολουθήσουμε εδώ τις εξελίξεις και θα συντάξουμε, θα συνεχίσουμε να συντάξουμε τις εκθέσεις. Όσον αφορά τώρα τη φορολογία, βεβαίως θα κάνω ό,τι μπορώ για να χρησιμοποιήσω τα εργαλεία της πολιτικής ανταγωνισμού για να αντιμετωπίσουμε και τις υποθέσεις όπου τα φορολογικά εργαλεία διευκόλυναν τον αθέμητο ανταγωνισμό. Όσον αφορά την ενέργεια, εδώ έχουν αληθεί πολλές ε, δεσμεύσεις ε, σε σχέση με την προσπάθεια ανοίγματος των αγορών. Ένα τελευταίο σημαντικό σημείο όσον αφορά μια ισορροπία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρών μελών, για παράδειγμα όσον αφορά το ενεργειακό μείγμα. Εδώ υπάρχουν κάποιες διαφορές όσον, υπά... Ε, όσον αφορά για παράδειγμα την πυρηνική ενέργεια. Αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μην διασπαθίζονται τα χρήματα των φορολογούμενων. Και πραγματικά σε ένα κοινοβούλιο που ενδιαφέρεται ε, πολύ για την ε, διαφάνεια. Θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια σχέση με τις ε, χρήσεις των χρημάτων των φορολογουμένων για να μπορούν ούτως ώστε να γίνονται και οι πολιτικοί εδώ υπόλογοι. Όσον αφορά την ψηφιακή ενιαία αγορά, η Επιτροπή αυτή πρόκειται να προωθήσει εδώ αυτές τις ε, προτάσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι για την εισφορά σας. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια πολύ καλή ε, πλατφόρμα για την ε, πολιτική ανταγωνισμού. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα το λόγο έχει ο εισηγητής κ. Μέσσερσμιτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για όλες αυτές τις παρατηρήσεις στη συζήτηση. Η πλειονότητα των σημείων πολιτικών και πολεμικών αναφέρθηκαν. Και θα ήθελα να αναφερθώ στο εξής. Μια εισήγηση είναι αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού. Και εδώ απευθύνομαι στους συναδέλφους μου Δανούς. Όταν υποβάλλουμε τροπολογίες είναι ο νόμος της πολιτικής ότι οι τροπολογίες μπορεί να αλλάξουν το νόημα της εισήγησης. Δεν μ' αρέσει εδώ οι δύο συνάδελφοι από τη Δανία που άρχισαν αυτήν την πολιτική, πολεμική και λένε ότι εγώ ε, άλλαξα, έκανα ε, άλλαξα τελείως και ότι δεν είμαι ο ίδιος. Όχι, χαίρομαι για το περιεχόμενο της εισήγησης. Η εισήγηση αναφέρει σημαντικά σημεία, κρίσιμα αλλά και επικοδομητικά. Παραδείγματος χάρη, τι χρειάζεται για να δημιουργηθεί μια εσωτερική ψηφιακή αγορά στο παρελθόν δεν ήμασταν τόσο ακριβείς, αλλά πρέπει να υπάρχει ε, διαλειτουργικότητα. Είναι σημεία που αναφέρουμε, είναι μια προοπτική ανάπτυξης. Αλλά αυτό συνεπάγεται η Κομισιόν αναλάβει πρωτοβουλία στην ψηφιακή αγορά και σε άλλους τομείς που αναφέρονται στην εισήγηση. Είναι θέμα εμπιστοσύνης, δέσμευσης, όπως ήδη το έχω πει. Πάντως να είστε βέβαιοι ότι θα ε, θα, έχουμε, θα είναι, είμαστε επικοδομητικοί αύριο σε αυτή την εργασία και εδώ απευθύνομαι σε αυτούς που έλαβαν το λόγο. Ναι, σε όλους δεν αρέσει πάντοτε ο συμβιβασμός, αλλά και εγώ καμιά φορά πρέπει να τον δεχθώ. Ένας συμβιβασμός δεν ικανοποιεί πλήρως ε, κανέναν, αλλά ε, γίνεται